να προχωρήσει στον δρόμο των φιλοδοξιών της να γίνει τμήμα της Ευρώπης. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε αυστηροί με αυτά που είμαστε στις εκλογές. Ευχαριστώ κύριε Ζαλεύσκη. Ο κύριος Σίδιετς για μισή λεπτό.